Καλησπέρα σας και κύριες και κύριοι. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, βλέπω και ιδίω οι βασικοί παίκτες της ομάδας ε, για την οδηγία για τις πληρωμές, οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Γνωρίζω βεβαίως ότι συνεχίζεται η η Εγώ έκανα έκκληση στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να βάλει ψηλά στην ατζέντα τα θέματα της εσωτερικής αγοράς και ελπίζω να συμφωνήσει και να έρθει και εδώ, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε στους ταινιστές, αλλά νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία εφόσον βρίσκεται σήμερα εδώ ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Για να συνεχίσουμε με, τις, με τα τυπικά. Έχετε ένα σχέδιο ημερήσιας διάταξης και αύριο θα βρισκόμαστε στην ίδια αίθουσα που είναι αρκετά μεγάλη και έχει και πολλή αντίχηση. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αύριο έχουμε και μία ενδιαφέρουσα έκθεση, την έκθεση BRICS και Grace, με συγχωρείτε, και επίσης θα έχουμε και την επιστροφή του καθηγητή, του κυρίου Μάριο Μόντι. Άρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ημέρα αύριο. Τώρα, σήμερα θα ασχοληθούμε με την έκθεση Βάιλερ και μετά θα περάσουμε στη συνάντηση των συντονιστών. Γιατί δυστυχώς ο κύριος Σαρκόφσκι δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, χρειάστηκε εκτάκτος να παραμείνει στην Πολωνία. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις. Απλά να σας πω και επισήμως ότι θα ήθελα παρακαλώ να εξετάσετε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων Φεβρουαρίου και Μαρτίου και αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις να μας ενημερώσετε μέχρι αύριο διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά και περνάμε σε μία από τις βασικές νομοθετικές εκθέσεις μας που βρίσκονται σε διαδικασία πρώτης ανάγνωσης υπό την κυρία Βάιλερ. Θα σας μιλήσει για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα σας πει και την άποψή της σχετικά και έχουμε εδώ και τους σκιώδεις συζητητές. Διόν είναι εδώ, ο κύριος Κοσνίσκι είναι ακόμη στην Ολομέλεια. Επίσης μετά μπορούμε να ακούσουμε και άλλα μέλη που ενδιαφέρονται για το λόγο. Η κυρία Μπρίκμαν είναι εδώ και ο κύριος Μπράιαντ που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ας ξεκινήσουμε όμως με την άποψη της κυρίας Βάιλερ για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ότι για μένα και πολλούς συναδέλφους ήταν αξιοπερίεργο ότι λάβαμε τόσες πολλές τροπολογίες και διαφορετικές θέσεις από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ενώ στην αρχή ε, είχαμε την εντύπωση ότι αυτό δεν πρόκειται να μας διευκολύνει, στην πραγματικότητα με συγχωρείτε, αλλά στα αγγλικά ακούμε πολωνικά. Θα ήθελα να ελεγχθεί το κανάλι. Λοιπόν, εγώ έχω ανοιχτό το μικρόφωνο μου. Με ακούτε τώρα? Λοιπόν, ε, ο, ο πρόεδρος τουλάχιστον πρέπει να με καταλαβαίνει, οπότε θα ξαναξεκινήσω. Οι πολλές τροπολογίες τις οποίες είχαμε ε, ξέπληξαν όχι μόνο εμένα αλλά και πολλούς άλλους. Από την άλλη πλευρά μπορώ ήδη να σας πω ότι είναι πολύ θετικό ότι πολλοί αντιφατικές απόψεις μπόρεσαν να συνδυαστούν σήμερα όταν είχαμε τη συζήτηση με τους Χιώδης και διαγράψαμε μία μία κεντρική γραμμή που θα χρειαστεί να ακολουθήσει η πορεία μας. Ε, καταρχήν όπως σας είπα χάρηκα διότι μέχρι αυτό το οποίο περιμέναμε και στηρίξαμε ε, με αυτή την νομοθεσία είναι κάτι το οποίο διατηρήσαμε και το μετατοπίσαμε κάπως από αυτό το οποίο επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αν ψηφίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα έχουμε soft law αλλά μη ένα βοήθημα και κυρώσεις. Νομίζω ότι θα υπάρξει μία νομοθεσία η οποία οποία δεν θα είναι ε, πάρα πολύ περίπλοκη, όχι με πάρα πολλές εξαιρέσεις και με μεγάλες διαφορές. Θα είναι μια νομοθεσία αντιθέτως η οποία θα ε, ισοσκελίσει τις ε, συναλλαγές στο δημόσιο και στις σχέσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Διότι στην ακρόαση φάνει ότι η πλειοψηφία αυτής της Επιτροπής είναι υπέρ μιας ενιαίας ρυθμίσεως με λίγες εξαιρέσεις. Δεν θα απαριθμίσω τώρα τις 200 τροπολογίες διότι η γραμμή την οποία ακολούθησαν οι σκιώδεις εισηγητές σήμερα το πρωί έδειχνε ότι θα μειωθούν πολλοί τροπολογίες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ανασκευασμένη οδηγία. Η συζήτηση και η διαπιστώση διαπιστώσεις ήταν πολύ χρήσιμες διότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπία. Καταρχήν όσον αφορά την ευκολία εφαρμογής και από την άλλη πλευρά διότι οι ρυθμίσεις που υπάρχουν ήδη σε ορισμένες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία ή οι κάτω χώρες θα μπορέσουν να συνεχίσουν να ισχύουν και σε ορισμένα σημεία πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία ε, ε, συμβιβαστική λύση. Νομίζω ότι ε, το βασικό είναι ότι όλοι οι σκιώδεις από όλες τις πολιτικές ομάδες που όλοι παρίσταντο σήμερα το πρωί μου είπαν σήμερα το πρωί ότι δεν θέλουν να υπάρξει μία εναρμόνιση μόνο όσον αφορά το ύψος των κυρώσεων δηλαδή το 2% ή το 1% για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά επίσης θα θέλανε να εναρμονίσουν και την προθεσμία καταβολής Οπότε μέχρι το τέλος Απριλίου νομίζω ότι παραμένει προς συζήτηση μόνο το θέμα των δημοσίων ε, συμβάσεων και αναθέσεων που πρέπει να, ε, να ρυθμιστεί. Ήταν δύσκολο για μένα να τα δεχτώ αυτά, δηλαδή 30 ημέρες πληρωμής ε, από το δημόσιο τομέα προς τον ιδιωτικό εκτός εξαιρέσεων που πρέπει να είναι αιτιολογημένες αυτό είχαμε ζητήσει από την αρχή και δεν μπορώ να είμαι τελεσίδικη γιατί θα ξανασυναντηθώ στην εβδομάδα του Στρασβούργου με τους Χιώδης αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε 60 ημέρες ε, προθεσμία καταβολής για τις, ε, ε, για τις συναλλαγές B2B μεταξύ ιδιωτών πράγμα το οποίο είναι μία απόκληση από την αρχική ε, ε, αρχή και ε, μας οδηγεί προς μεγαλύτερη εναρμόνιση και εγώ προσωπικά και όχι μόνο εγώ προσωπικά αλλά και η πολιτική μου ομάδα η οποία με στήριξε στην ε, πολιτική διατύπωση ε, ότι η ελευθερία των επαφών και των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διατηρηθεί ε, και πιστεύω ότι στην Επιτροπή αυτή η πλειοψηφία ε, θέλει να τονίσει περισσότερο την εναρμόνιση παρά την ελευθερία του συμβάλλεστε, freedom of contract και ε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό αναφέρεται εις ε, την ε, ομάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις οποίες θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτές τις συναλλαγές διότι ένα μέρος αυτού του κύκλου ήθελε περισσότερη ευελιξία και το άλλο περισσότερα αυστηρότηση. Αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι δεν μπορούμε όλους να τους ικανοποιήσουμε και ως εκ τούτου θα διατυπώσω και θα στηρίξω την πρόταση να υπάρξει μία ρύθμιση ε, B προς B με μία συμβιβαστική πρόταση καταβολής εντός 60 ημερών και θα το υποβάλω προς ψηφοφορία. Ε, αυτές είναι οι γενικές γραμμές. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θέματα για το πώς θα ρυθμίσουμε, ε, πώς ε, θα, πού θα τοποθετήσουμε και πώς θα διαμορφώσουμε το πέναλτι, το οποίο δεν θα είναι μία τιμωρία αλλά μία αύξηση του, των επιτοκίων, ε, θα οδηγήσουν σε μία έκβαση η οποία δεν με προβληματίζει και πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη δεν είχε διαγραφεί τόσο σαφώς στην τελευταία τελευταία προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε διότι η ομάδα ζητούσε μία εναρμόνιση και αυτό επιθυμούσαν και οι συνάδελφοι των συντονιστών αλλά και τα μέλη της Επιτροπής που δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, πολύ εκτενή παρουσίασή σας και ε, θα ε, εστιαστούμε σε ορισμένα θέματα όσο θα συζητάμε αλλά αντελήφθηκα ότι έχετε συμβιβασικές τροπολογίες για τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί και θα διευκολύνουν πολύ τη δουλειά μας. Η κυρία Χάνσλικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια διότι η συνεργασία υπήρξε εξαιρετική και πολύ θετική μέχρι τούδε και η συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί μεταξύ οδών συντονιστών συνέβαλε στην καλή συνεργασία. Όσον αφορά την θέση της πολιτικής μας ομάδας, όντως έχουμε υποβάλει μία σειρά από τροπολογίες οι οποίες τροπολογίες μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερα σημεία αλλά από το προχωρήσω θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου στο θέμα των ε, καθυστερημένων πληρωμών δεν πρέπει να αναφερθούμε μόνο στις δημόσιες συμβάσεις αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να προσπαθήσουμε να τις διευκολύνουμε εις την εσωτερική αγορά και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η οδηγία για τις καθυστερημένες ε, πληρωμές σε εμπορικές συναλλαγές θα είναι θετική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα τις βοηθήσει διότι μόνο όταν θα έχουμε ρυθμίσει το θέμα αυτό θα μπορέσουμε να μιλάμε για μια αποδοτική και λειτουργική εσωτερική αγορά όταν ήδη οι κανόνες θα ισχύουν για όλους. Γιατί αν σε μια περίοδο κρίσεως θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ρευστότητα ενδιαφέρει αυτές τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πληρώνονται αυτά τα οποία τους χρωστούνται εγκαίρως. Και γι' αυτό αυτό στις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει ζητούμε μία εναρμόνιση ε, και σε επίπεδο σχέσεων ε, β προς β, δηλαδή μεταξύ δύο εταιριών. Ε, δηλαδή στις συμβάσεις αυτές θα θέλαμε να υπάρχει ε, ως ανώτατο περιθώριο πληρωμής η περίοδος των 60 ημερών. Όσον αφορά τις ε, δημόσιες αρχές και τον, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπάρχει, έχουμε συμφωνήσει σε κανόνα 30 ημερών συν επιπλέον 30 εάν υπάρχουν ιδιάζου σε συνθήκες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η τιμωρία, οι κυρώσει σε αυτό το θέμα δεν θα οδηγήσει υποχρεωτικά σε θετικά αποτελέσματα και αναφέρουμε εδώ στην πρόταση του 5%. Το βάρος αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τις εταιρείε. Και όταν μιλάμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις γενικότερα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν απαιτούν επιπλέον κυρώσεις και ανταμοιβή ε, οι επιχειρήσεις αυτές απλούστατα να πληρώνονται στο συμπεφωνημένο χρόνο και ε, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ε, απορρίψουμε την πρόταση του 5% και οι περισσότερες ακούν ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση και όπως είπε και η κυρία Βάιλαρ σήμερα μετά τη σημερινή συνάντηση καταλήξαμε σε μία συμφωνία και μάλλον θα διαγραφεί η πρόταση του 5%. Τώρα, όσον αφορά τα διάφορα άλλα τέλη, συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές πρέπει να την χάνουν τις ίδιες μεταχειρήσεων. Ορισμένες ε, ε, από τις τροπολογίες είναι καλές αλλά ελπίζω θα καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση. Εγώ θα είμαι υπέρ ε, ενός, ε, ενός ε, ποσού 100 ευρώ άλλοι όμως ζητούν να μην υπάρχει κατά το 100 ευρώ αλλά ένα ποσοστιαίο μια ποσοστιαία καταβολή και αυτά είχα να να πω και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς βλέποντας τα πράγματα έτσι, αυτό που κάναμε και αυτό είναι μια έκπληξη, βρήκαμε ένα συμβιβασμό που εγκρίθηκε ήδη που στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τίνει χείρα βοηθείας. Βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός ήταν ο στόχος. Και αυτό απαιτεί και αλλαγή νοοτροπίας του συστήματος. Φυσικά δεν μπορεί κανεί με ένα σύμβασμο να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες πρότεινε 5% σε σχέση με τις κυρώσεις επιτροπή. Μετά υπήρξε συζήτηση αν θα είναι εντάξει να έχουμε μόνο τις ε, κρατικές ε, και όχι τις ιδιωτικές ε, υποθέσεις και το θέμα της ίσης μεταχείρισης είναι ένα ζήτημα. Το αναγνωρίζουμε και σε σχέση με τις κυρώσεις αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Στο δικό μας σύστημα το νομικό δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρόστιμα και για το σύστημα αυτό και τη συζήτηση για αλλαγή συστήματος που έγινε συζήτηση, αλλά κυρίως για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το είπε η συνάδελφος Βάιλερ, είναι απλούστερο σε σχέση με τις ρυθμίσεις της Επιτροπής. Είναι πολύ απλό και ουσιαστικά μπορεί με τρεις προτάσεις να επεξηγηθεί. Έχουμε ελευθερία του συμβάλλεστε με 30 ημέρες προθεσμία που μπορεί να επεκταθεί σε 60 ημέρες. Μετά ελευθερία του συμβάλλεστε στις ιδιωτικές υποθέσεις μέχρι 60 ημέρες μπορούν να συμφωνήσουν ε, μέσα στο πλαίσιο αυτό αλλά όχι πέρα από αυτό. Σε όλες οι συζήτησεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας έλεγαν πάντα ότι περισσότερο θα βοηθούσε αυτό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι ένα, μια νομική υποχρέωση σε σχέση με τέτοιες πληρωμές ε, πέρα από τις 60 ημέρες δεν θα και αυτό θα βοηθούσε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό είναι όλο και όλο. Δεν χρειάζονται περισσότερε εξηγήσει και υπάρχει και συνένεση για την ανάκτηση κονδυλίων, recovery costs, να μην υπάρχει δηλαδή υπερβολική γραφειοκρατία. Τη μία ή άλλη λεπτομέρεια μπορούμε να τις ε, διευθετήσουμε. Πρόκειται για αλλαγή υποδείγματο και προτύπου σε σχέση με τι 60 ημέρε και σε σχέση με ε, πρόστιμο το οποίο θα επεβάλλεται με, τις, ε, με τους τόκους που θα ανέβαινε σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής στο 9%. Και αυτό αντικαθιστά φυσικά τις ε, πληρωμές ε, κυρώσεων σε σχέση με το 5% που είχε προταθεί. Είμαστε στη συνάντηση που είχε γίνει σε σχέση με τους κοιόδης. Θα ξανασυναντηθούμε στο Στρασβούργο, θα δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και τέλη Απριλίου θα ληφθεί απόφαση από αυτού. Ευχαριστώ. Uh, θα σε ευχαριστώ κυρία Ρούλε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Θα ήθελα όμως ένα σημείο να αναφέρω που εγώ από πλευράς διατύπωσης έχω κάποια αντίρρηση σε σχέση με αυτά. Το θεωρώ σημαντικό να μην κάνουμε λόγο για τιμωρίες και ποινές και πρόστιμα. Αυτό που θέλουμε είναι σε περίπτωση καθυστερήσεων να αυξάνονται τα ε, επιτόκια, να, αυξάν, να αυξάνονται με συγχωρείτε οι τόκοι. Αυτό δεν είναι ε, τιμωρία, αλλά είναι ε, λόγω καθυστερημένης πληρωμής, λόγω καθυστερημένης εξόφλησης αυξημένο ποσό το οποίο καταβάλλεται. Και σωστό αναφέρθηκε από τον κύριο Κρότσμαν ότι σε σχέση με την ε, αντικατάσταση της ε, πίνης ε, θα γίνεται μόνο λόγος για καθυστερημένες πληρωμές ε, και με αυξημένους τόκους. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο θα μπορούσαμε εμείς να συμφωνήσουμε ως ομάδα. Για να μην υπησέρθουν πάλι, μην παρισφρέουν εδώ οι έννοιες της τιμωρίας ή της ποινή. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα απορρίψουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. And then finally from uh, shadows, Mr. Uh, and then... Τέλος, και μετά τους σκιώδεις έχουμε Γκέπχαρτ, Ιντάλγο, Μπουζόη και Βανιόλ. Αν υπάρχει και άλλος που ενδιαφέρεται, παρακαλώ να μας ενημερώσει. Ο κύριος Διόγκ προς το παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους συγχάρηγαν ήδη την κυρία Βάιλερ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω τα συγχαρητήρια εκ μέρους των σκιωδών ισογητών. Ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία μαζί της και ο τρόπος με τον οποίο εξετελέσθη. και εγώ από την πλευρά μου είμαι αποφασισμένος να υπάρξει απλοποίηση των τροπολογιών. Για παράδειγμα, έχω κάνει μια τροπολογία για τα business to business προκειμένου να μειωθούν στα 30 στις 30 ημέρες, αν και από ό,τι φαίνεται προτιμούν κάποιοι τις 60 ημέρες, γι' αυτό θα συμβιβαστώ. όσον αφορά την αύξηση των ποσοστών επιτοκίων θα συμφωνήσω και εδώ με την πλειοψηφία προκειμένου να υπάρξει συνένεση. Τώρα όσον αφορά την ελευθερία σύναψης συμβάσεων. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη ελευθερία στο θέμα των συμβάσεων. Ήδη υπάρχουν πολλές θέμητες πρακτικές και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσφύγουν στα δικαστήρια για παραβίαση των όρων των συμβάσεων. Αυτό υπάρχει ήδη στην πράξη λοιπόν, αλλά αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να έχουμε πιο σαφή κριτήρια προκειμένου να μην αυξηθούν πολύ οι διάφορες αντιδικίες. Τώρα, κάτι όπου δεν θα συμφωνήσω με τους υπολείπους όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τις δημόσιες αρχές στις κάτω χώρες πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες υπερβαίνουν αυτή την προθεσμία των 30 ημερών. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δώσουμε εξαίρεση θα υπάρξουν πολλά προβλήματα. Αν θέλετε να αλλάξουμε την προθεσμία καλώς, αλλά να μην έχουμε πολλές εξαιρέσεις που απλά θα αυξήσουν την πολυνομία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Χουάνιοκ και σφά επίσης έχουν ζητήσει το λόγο. Όμως πρώτα η κυρία Γκέπαρτ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και να ευχαριστήσω και την Μπάμπα Βάιλερ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και που δεν είναι καθόλου απλό θέμα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πρόκειται για τους όρους ε, ε, λειτουργίας ε, των εταιριών, επιχειρήσεων ιδιωτικών και κρατικών και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Κατά τούτο λοιπόν βρισκόμαστε σε καλή οδό, σε καλή πορεία να έχουμε μια καλή έκθεση που θα εγκρίνουμε υπερψηφίζοντα την. Και από όλε τι κοινοβουλευτικέ ομάδε, όπω άκουσα μέχρι τώρα, μπορεί να υποστηριχθεί, θα υποστηριχθεί και αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Παρ' όλα αυτά όμω πρέπει κάπω να, εκφράσω, να εκφράσω την έκπληξή μου για την εξέλιξη των συζητήσεων που έγιναν. Και πρέπει την Μπάρμπαρα Βάιλερ, μια και και εκείνη θα εξεπλάγει το ότι ξαφνικά τώρα θα πρέπει κάποια πράγματα εδώ να ενταθούν. Παρότι σε όλες οι συζητήσεις μέχρι τώρα όταν επρόκειτο για κάποια θέματα που επρόκειτο για ελευθερία του συμβάλλεστε, συμβατική ελευθερία, είχαμε την αντίθετη θέση. Η δεξιοί ήταν εκείνη μέχρι τούδε που πάντα είχαν εγγράψει στις σημαίες τους το θέμα της ελευθερίας του συμβάλλεστε και εμείς είμαστε εκείνοι που θέλαμε να έχουμε περισσότερες ρυθμίσεις και τώρα τα πράγματα φαίνεται να έχουν αντιστραφεί. Μπορούμε όμως να δεχτούμε έστω και κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όμως στην ομάδα μου. Να δούμε αν υπάρχει συνένεση, συνενετική θέση για αυτή, αυτό το συμβιβασμό. Όμω θέλουμε ως ομάδα να μην δημιουργήσουμε με κανένα τρόπο προσκόμματα και εμπόδια. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα. Όμω ω προς αυτό θα ήθελα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Νομική Υπηρεσία για αυτό το θέμα να ακούσω ποιε απόψει έχουν διότι έχω την, το φόβο ότι αν εμείς σε ένα τέτοιο τομέα πάμε υπερβολικά μακριά όπως με μια τέτοια πρόταση και με τον ε, το θέμα της ελευθερίας ε, του συμβάλλεστε και όταν λέτε εσείς κύριε Κρόσμα σε 60 ημέρες ε, θα υπάρχει αυτή η ελευθερία μέσα σε αυτά τα πλαίσια Μήπως αυτό θα οδηγούσε στο να μην υπάρχουν πλέον κάποιες ρυθμίσεις επειδή το Συμβούλιο δεν θα ακολουθούσε μια τέτοια θέση. Θα έλεγε ίσως αυτό είναι απαράδεκτο για μας. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Να μην χρησιμοποιηθεί αυτός μοχλός για άσκηση πίεσης και στο τέλος να μην έχουμε καμιά ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο και έχουμε ανάγκη να ακούσουμε πώς τοποθετούνται τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέπχαρτ και εγώ ως πρόεδρος αλλά και η γραμματεία όντως θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις είναι νομικώς ορθές και θα το συζητήσουμε αυτό και με τη γραμματεία γιατί πρέπει να το γνωρίζει αυτό η Επιτροπή πριν την ψηφοφορία. Ο κύριος Συντάλγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ εσάς Πρόεδρε για την ικανότητά σας την νομική και την κοινοβουλευτική ώστε σε αυτή την Επιτροπή να έχει προχωρήσει, να έχει πάρει αυτή την οδηγία όταν στην νομική επιτροπή υπήρχε αγώνας ώστε το σύνολο αυτής της οδηγίας ε, να την εκπονούσαμε εμείς ε, και το ξέρετε χάσαμε όμως. Ε. Όμως προσέξτε, προσέξτε το είπατε εσείς, το είπε και η Εύελιν πιο πριν, το γεγονός ότι, συγγνώμη, υπάρχει τρομερή παρέμβαση στο μικρόφωνο σας, μικροφωνισμός. Ίσως θα μπορούσατε να μετακινηθείτε σε ένα άλλο μικρόφωνο ίσως. Γίνεται αυτό, μπορείτε να μετακινηθείτε σε άλλη συσκευή. Ωραία, για να το δούμε. Ah, ah, ah. Εντάξει, συγγνώμη. Είχα το κινητό μου. Η κίνησή μου δεν είναι και πολύ εύκολο να φτάσω σε άλλο. Τέλος πάντων έλεγα όμως ότι το γεγονός ότι όπως πολύ καλά είχατε πει, ότι πρέπει να νομοθετήσουμε σωστά. Άκουσα στη συζήτηση ότι <clears throat> να ως μάνα εξ ουρανού επιχειρήσεις να καταλήξουμε σε αυτή την οδηγία στις εργασίες μας. Το πιο σημαντικό είναι ως νομοθέτες να νομοθετούμε σωστά και καλά και να νομοθετούμε με βάση το δίκαιο και ευθυγραμμιζόμενοι προς τις ανάγκες του δικαίου. Και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που ανήκω ως πλήρες μέλος σε προσπαθήσαμε σε σχέση με ένα ή άλλο θέμα, ε, ένα ή άλλο άρθρο, αλλά προσπαθήσαμε και με τροπολογίες να ε, προχωρήσουμε. Μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση στο ότι στη συζήτηση σήμερα βρισκόμαστε σε κάποιες ε, θέσεις που ε, η κατάργηση των ε, κυρώσεων στο άρθρο 5 σε σχέση με το απαράδεκτο που είχε παρουσιαστεί όσον αφορά το, την καλή νομοθεσία. Χαίρομαι λοιπόν ότι στο τέλος καταλήξαμε στις κοινοβουλευτικές εργασίες ώστε να είμαστε σε σωστή θέση. Όμως παρισφρέουν κάποιες τροπολογίες εδώ και κάποιες θέσεις που δίνουν κάποιες ε, μη τυπικές κυρώσεις ε, που θα έπρεπε και αυτές να απορριφθούν. Αναφέρομαι στον Ισπανό συνάδελφό μου και πολύ καλό φίλο μου τον κύριο Τσεβαρία όταν λέει ο κύριος Ετσεβαρία ότι ένας τρόπος για να καταπολεμήσουμε αυτά τα πράγματα είναι να εισαγάγουμε μια ασφάλεια, μια ρήτρα ασφάλειας ότι στις πέντε επόμενες ημέρες μη πληρωμής από, από επιχειρήσεις να υπάρξει μια ρήτρα ασφάλειας που θα αναλαμβάνει να πληρώσει αυτές τις ε, οφειλές. Αν υπάρχει προηγούμενη ασφάλεια, εντάξει. Αν όμως μια εκ των υστέρων ασφάλεια σε σχέση με αυτές τις πέντε ημέρες, δεν θα ήταν σωστό αυτό. Και όσον αφορά την απόλυτη ανεξαρτησία, όσον αφορά τον ε, συνάδελφό μου ε, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, θα, αν δεν πίστευα σε αυτή του την ακαιρεότητα, θα πίστευα ότι κάποιοι λομπιίστες θέλουν εδώ να προτείνουν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε υπερβολική δαπανηρή ε, διαμόρφωση της οικονομικής μας ζωής και δεν θα ήταν σωστό για αυτήν την οδηγία. Όσον αφορά τα, τους τόκους ε, για την καθυστέρηση θα πρέπει να περιορίζεται στο νόμιμο τόκο. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος ορισμός πέρα από το νόμιμο τόκο διότι σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να βλέπαμε ότι μεγάλες επιχειρήσεις θα είχαν σε σχέση με, τα, ε, με τους τόκους ε, θα μπορούσαν να διαμορφώσουν διαφορετικά πλαίσια για, το, για λογαριασμό τους. Δεν είναι λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Να δώσουμε χείρα βοηθεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην επιβαρυνθούν σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Να μην χρειάζεται δηλαδή να ε, δεχθούν μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πράγμα το οποίο θα ήταν αντίθετο με με, το, με την πρόθεση του νομοθέτη που θα θέλαμε να ε, είμαστε σωστοί. Και τέλος θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, ότι επίσης υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, η διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής της οδηγίας όσον αφορά τον, τη δημόσια υπηρεσία ή τις δημόσιες υπηρεσίες. Η κυρία Μούνιθ και εγώ και σε σχέση με τις τροπολογίες ε, είχαμε μια πολύ περιοριστική, ας το πούμε έτσι, ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο σε σχέση με τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, ε, σε σχέση με την προστασία πληρωμών. Διότι αν εισάγουμε εδώ το ότι οι επιχειρήσεις με δημόσιο κεφάλαιο ή με δημόσιο ε, ε, με πλειοψηφία του δημοσίου ε, σε αυτές. Αν ρυθμίζαμε ξεχωριστά αυτές θα ήταν πολύ μεγάλος κίνδυνος. Το να δούμε ότι εδώ οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να έχουν ένα ξεχωριστό πλαίσιο ε, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει να δούμε τους περιορισμούς που δημιουργούνται για την καλή λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων που τις αποκαλούμε δημοσίου συμφέροντος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν νομίζω παρά να έχουμε ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο, πολύ περιορισμένο πλαίσιο για την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας ή δημοσίου ωφέλους. Γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε καλοί νομοθέτες και δεν θα είμαστε σωστοί και δεν θα είμαστε σωστοί όσον αφορά το έργο μας να είμαστε αρμόδιοι και να ρυθμίσουμε σωστά το πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας ε, και μας εκθέσατε τις απόψεις σας. Είστε ευπρόσδεκτος και στο μέλλον. Συνεχίζω όμως με Μπενζόη, Βανιόη και τα λοιπά. Θα ήθελα να κλείσουμε εδώ την λίστα για να μην καθυστερήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Αν και βεβαίως δεν θέλω να σας πιέσω γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Κύριος Πεζόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση που συζητούμε πραγματικά είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι εκείνοι που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα πρέπει να υποχρεούνται να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους κυρίως όταν πρόκειται και για δημόσιες υπηρεσίες όταν υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών καθυστέρηση πληρωμών τροχοπεδούν τη δραστηριότητα για παράδειγμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσχεραίνουν και την οικονομική κατάσταση εφόσον τροχοπεδείται η δραστηριότητά τους στα κράτη-μέλη. Θέλω να χαιρετήσω τη δραστηριότητα της κυρίας Βάιλερ και του σκιώδου συζητητού κ. Κρότσμαν. Με τον ένα ή άλλο τρόπο κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβασμούς. Όσον αφορά τις πιο σημαντικές πτυχές, τις ουσιοδέστερες πτυχές αυτής της πρότασης θα έλεγα όμως ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε περισσότερο αυτό το 5% όσον αφορά την κύρωση ή το πρόστιμο να το διατηρήσουμε όχι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Ένα μέρος των φιλελευθέρων συμφωνούν με αυτή την άποψη γιατί διαφορετικά θα, η, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα την καθιστούσαμε αρκετά αυστηρή όταν έχουμε προθεσμία 30 και 60 ημερών για τις ε, πληρωμές, τι θα γίνει αν και η προθεσμία των 60 ημερών δεν θα τηρείται πού θα οδηγηθούμε. Αν δεν υπάρχει λοιπόν πραγματική δυνατότητα να υπάρχει κύρωση ή πρόστιμο, τότε πολλά κράτη-μέλη αυτή την οδηγία δεν θα, την εφαρμο... δεν θα θέλουν να την θέσουν σε εφαρμογή. Αυτό που εμείς συζητήσαμε ως συμβιβαστική λύση νομίζω θα τύχει υποστήριξη από όλους και ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ προστίθεται και νέοι στην λίστα. Παρακαλώ, αν θέλετε κι εσείς να προσθεθείτε, ενημερώστε μας. Η κυρία Ρόιτεβα ήταν η τελευταία που προσθέθηκε. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα Βάιλερ για τον χρόνο που έχει αφιερώσει, για τις πολλές συναντήσεις που είχε με όλους τους φορείς. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για σημαντικό θέμα και έχω και εγώ, όπως και πολλοί συνάδελφοι, ανησυχίες για τις διακρίσεις που κάνει η Κομισιόν μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων Επίσης, ε, όπως και ο κύριος Χουάνγκ σκέφτομαι ότι ίσως θα ήταν απλούστερο να διαγραφεί το άρθρο 5 και να παραμείνει ένα άρθρο 3 που θα καλύπτει τους πάντες ανεξαρτήτως καθεστώτος. Βλέπω ότι και άλλες πολιτικές ομάδες σκέφτηκαν κατά τον ίδιο τρόπο, μόνο που αυτοί διέγραψαν το άρθρο 3 και προσάρμοσαν το άρθρο 5 το βασικό είναι να περάσει αυτή η ιδέα. Επίσης υπάρχει κάποια διάταξη συγκεκριμένη για τις 60 ημέρες όσον αφορά το νοσοκομιακό σύστημα, γιατί εκεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συστήματος υγείας. Σε ορισμένες χώρες είναι πραγματικά αδύνατο να γίνει σεβαστή αυτή η προθεσμία των 30 ημερών εκεί, χωρίς να υπάρξει υποψία για κακή πρόθεση. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να επιτρέπει τις καταχρηστικές καθυστερήσεις πέρα από τις 30 ημέρες. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ποινές από την πρώτη μέρα της καθυστέρησης μετά το πέρας της προθεσμίας γιατί κάτι τέτοιο θα ίσχυε θα σήμαινε διπλή ποινή εφόσον υπάρχουν και τα οι προσαυξήσεις για τις καθυστερήσεις. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η Μπάρμπαρα Βάιλερ σίγουρα θα προσπαθήσει να βρει τους κατάλληλους συμβιβασμούς που θα είναι και επικοδομητικοί και θα βελτιώσουν το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Μπάρμπαρα για την ποιότητα του έργου της ε, και για τους σκόπους ε, που έκανε. Η Μπερναντέτ ε, με κάλυψε αρκετά γιατί είχαμε συζητήσει αυτά τα θέματα και είχαμε συντονιστεί στο θέμα των τροπολογιών, ειδικά όσον αφορά τις οι δημόσιες υπηρεσίες. Να προσθέσω λοιπόν μόνο κάτι. Όσον αφορά τις ε, τα πρόστιμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που να μπορεί όντως να αποτρέπει. Για αυτό το λόγο προτείνουμε 3% για καθυστέρηση πέρα των 60 ημερών και 5% για καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν αρκετά επικοδομητικό προκειμένου να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις. Αυτά. Κύριε Σβάμπ. Θα είμαι σύντομος διότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις ε, που έγιναν πιο πριν και για τις επικοδομητικές παρεμβάσεις ε, από πλευράς κυρίας Βάιλερ θέλω να ευχαριστήσω. Νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εξής. Το impact assessment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε σαφώς ότι ο αποφασιστικός παράγοντας για την υλοποίηση καθυστερημένων πληρωμών είναι η λήψη υπόψη σε σχέση με υφιστάμενες εργασιακές ή συμβατικές επαφές. Και κάτι τέτοιο σε σχέση με τη ρύθμιση δεν θα άλλαζε. Ναι, μεν το θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών με καθαρό τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί με τον ε, συμβιβασμό αλλά το πρόβλημα, τα αιτήματα αυτά να μην περνάνε από πλευρά επιχειρήσεων δεν επιλύονται. Δεν επιλύονται στη ρίζα του ή στη βάση τους οι καθυστερήσεις. Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι 60 μέρες ίσως θα ήταν υπερβολικά σκληρή η ρύθμιση και έχουμε και το θέμα της μη ύπαρξης ρύθμισης. Σήμερα έχουμε τη ρύθμιση 30 ημερών και 7% τόκων για την καθυστέρηση. Έχουμε κάτι λοιπόν. Αν δεν είναι πρόθυμο το Συμβούλιο να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρό όλα τα ε, ανεπίλητα, τα μη ε, λιμένα προβλήματα, τότε μπορούμε να δούμε ότι σε σχέση με την ε, μη ρύθμιση από πλευρά των κρατών μελών, τότε θα ήταν ίσως ε, κρίμα για τη δουλειά που έχουν κάνει ε, οι συγγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές, αλλά δεν θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας εμείς. Τώρα, με το 9% η τόκη είναι ε, σχετικά υψηλή, πρέπει να το πούμε. Και όταν υπάρχει εδώ το αίτημα αποζημίωσης και όταν υπάρχει και τεκμηρίωση για νόμιμη αποζημίωση, μπορεί το ποσό αυτό να είναι ακόμα, πιο, ακόμα μεγαλύτερο. Και εν τέλει θα ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος πιο πριν. Νομίζω με τη δική μας πρόταση και εγώ δεν είμαι φυσικά εκπρόσωπο μια δεξιά ε, κοινοβουλευτική ομάδα όπω εσεί είπατε. Δεν είμαι δεξιό. Είμαστε εμεί ε, στο πολιτικό κέντρο βρισκόμαστε. Και σε σχέση τώρα με τη γενική ρύθμιση, το 60, 60 ημέρε ω ανώτατη ρύθμιση μπορεί να ε, γίνει δεκτή και έτσι επιλύουμε τα προβλήματά μα. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Mrs. Νομίζω ότι, ελπίζω ότι εκπροσωπώ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι ολόκληρη η ιδέα αυτού του κανονισμού είναι ακριβώς να μειώσει τη γραφειοκρατία, να αποφύγει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά το στόχο, ελπίζω να μην με παρανοήσετε, αλλά στο πρώτο άρθρο λέγεται ότι θα αναφερόμαστε σε όλες τις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές και στη συνέχεια λέγεται ε, από ε, οικονομικούς φόρους ε, φορείς προς άλλους οικονομικούς φορείς ή μεταξύ οικονομικών φορέων. Δηλαδή εγώ θεωρούσα από την αρχή ότι οι σχέσεις Β προς Β ήταν ένα ουσιαστικό μέρος αυτής της νομοθεσίας ε, διότι οι μικρές ε, εταιρείε δεν πληρώνονται και από άλλες εταιρείε, όχι μόνο από το δημόσιο. Επίσης δεν υπάρχουν μόνο πιστωτές υπάρχουν και χρεώστες και είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να κοιτάξουμε. Βεβαίως ε, συγχαίρω τη Μπάρμπαρα, ευχαριστώ τους πάντες, όλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά, αλλά αφού ευχαριστήσω θέλω να πω και μερικά σχόλια, διότι είδα ότι σε περίοδο κρίσεως η ελευθερία του, ε, των ε, συμβάσεων είναι πολύ βασική και γι' αυτό προσπαθούμε να καταρτήσουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο για να αποφύγουμε και χρεοκοπίες, να αποφύγουμε προβλήματα. Θα ήθελα ακόμη και η φίλη μου δίπλα μου να ε, μπορεί να εξετάσει ε, το θέμα της ελευθερίας των συμβαλωμένων να συμφωνήσουν σε 90 ημέρες διότι υπάρχουν τομείς όπου η διαφορά αυτή μπορεί να είναι μία εξαίρεση αλλά μπορεί να δώσει μια ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία εξαίρεση για τις μεγάλες, για τις δημόσιες αρχές. Διότι οι ιδιώτες αναλαμβάνουν κινδύνουν. Αλλά το, το δημόσιο έχει γραμμές προπολογισμού που κάποιος έχει αποφασίσει. Και απλώς υπάρχει γραφειοκρατική η καθυστέρηση, δεν λειτουργεί το σύστημα και δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ε, προσχήματα για να τιμωρούμε περισσότερο τις εταιρείες. Όσον αφορά, τις, ε, όσον αφορά τις χειρώσεις, θα, θα αφαιρούσα τα ποσά κατά αποκοπήν και θα έπαιρνα μόνο μία αύξηση ποσοστιαία. Δεν είναι σωστό να έχει ε, κανείς ε, κατά αποκοπήν ποσά ε, διότι διαφορετικά εφόσον ο στόχος της κυρώσεως είναι να καλύψουμε τα έξοδα που έγιναν θα πρέπει αυτά τα έξοδα να αποπληρώνονται και αυτό είναι ε, κάτι που δεν μπορούμε να καθορίσουμε εκ προημίου, απλώς θέλουμε όντως να υπάρχει πληρωμή και σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άριας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια για αυτό το έγγραφο, την κυρία Βάιρερ. Έκανε πραγματικά καλή δουλειά ανεξάρτητα από τις παρεκκλήσεις απόψεων που είχαμε πολλοί από εμάς σε σχέση με το αρχικό κείμενο και με την ικανότητα αυτού του εγγράφου, αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας να επιλύσει πραγματικά το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών όσον αφορά τις διάφορες επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντος όμως είμαι βέβαιος ότι και το έγγραφο αλλά και οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν μόνο ως αντικείμενο την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται και που όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις πληρωμών. Θα ήθελα να πω στον συνάδελφο πιο πριν ότι στην τροπολογία που ανέφερε δεν κάνω λόγο για ασφάλεια, κάνω λόγο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η ιδέα για την ασφάλεια που αναφέρθηκε θα μπορούσε να είναι και καλή κιόλα. Όχι να συμπεριληφθεί εδώ στο νομοθετικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας, αλλά θα ήταν μια καλή ιδέα, ώστε να μπορέσουν οι δύο συμβαλόμενοι όταν υπογράφουν μια τέτοια σύμβαση να το λάβουν υπόψη. Θα μπορούσε να είναι κάτι που ε, κατ' επιλογή θα μπορούσαν να κάνουν. Τώρα, σε σχέση με την ε, τροπολογία μου, αποστεριόρι είναι εκ των υστέρων, διότι πιστεύω ότι είναι καλές οι προθέσεις ε, της δημόσιας υπηρεσίας ε, όταν ε, υπάρχει μια τέτοια σύμβαση που συνάπτεται με μια τέτοια δημόσια υπηρεσία. Το πρόβλημα δεν είναι το, η, η υπογραφή μιας σύμβασης, το αντίθετο όταν υπάρχει υπογραφή μια σύμβαση ε, για μια επιχείρηση αυτό είναι ε, λόγος ικανοποίησης. Το πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα, όταν δεν πληρώνονται οι εργασίες ή δεν καταβάλλονται τα χρεωστούμενα. Ε, Πιστεύοντα πάντα στι καλές προθέσεις των συμβαλωμένων. Αυτή λοιπόν η ιδέα έχει ως ιδέα να επιλύσει το πρόβλημα το οποίο τίθεται και να το επιλύσει με ταχύ τρόπο και υπεύθυνο τρόπο. Είναι ακριβώ ε, η ίδια πρόθεση που υπάρχει κατά την υπογραφή μια σύμβασης. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για τιμωρία ή κύρωση θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για κύρωση ή ποινή μόνο αν η δημόσια υπηρεσία δεν υλοποιεί, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρότεβα και μετά ο κύριος Άγγος, ο οποίος ε, έφτασε καθυστερημένος αλλά θα έχει σαν σοβαρό ε, λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα <clears throat> να χρησιμοποιήσω το χρόνο για να αιτιολογήσω τις τροπολογίες μου. Πρόκειται για έναν κανονισμό και πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς όσον αφορά την ε, διατύπωση. Γι' αυτό ε, και έχω προτείνει μια τροπολογία στο άρθρο 4, διότι εδώ πρόκειται για συσσωρευτικούς λογαριασμούς, διότι παραδείγμα χάρη θα ήθελα να σας πω ότι ένα νοσοκομείο έχει, έχει παραγγείλει παραγγέλνει από κάποιον προμηθευτή ένα φάρμακο και επαναλαμβάνει πολλές τέτοιες, τέτοιες παραγγελίες μέσα στην ίδια ημέρα και μπορεί να δημιουργηθούν πολλοί λογαριασμοί. Οπότε Οπότε εάν ε, αυτό επαναλαμβάνεται μπορεί να θεωρηθεί ε, σαν, μία, ε, σαν ένας συσσωρευτικός ο λογαριασμός του. Συζήτησα λοιπόν με νομικούς εμπειρογνώμονες και ε, για να αποφύγουμε ε, να ε, έχουμε διάφορα τιμολόγια τα οποία είναι βολιδοσκοπιστικά και να έχουμε ένα τελεσίδικο λογαριασμό θα πρέπει να διαχωρίσει κανείς τις κυρώσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων και να διευκρινίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Στο άρθρο 5, το άρθρο 5 θα έπρεπε να καταργηθεί όπου μιλάμε για τις, ε, ε, για τις κυρώσεις 5% προς το δημόσιο. Επίσης θα ήθελα να καταργήσουμε και τις 60 μέρες διότι πιστεύω ότι αν η προθεσμία αυτή δεν είναι σωστή τι θα εφαρμόσουμε. Εμείς κοιτάμε να απλοποιήσουμε και τις κυρώσεις, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι κατά αυτόν τον τρόπο οι, οι, οι, καθυστερημένες πληρωμές θα εκτελούνται πιο γρήγορα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικές συνθήκες για το δημόσιο και διαφορετικές για τους ιδιωτικού συναλλασσόμενους διότι κάθε χώρα θα μπορούσε να καθορίσει τι θεωρεί ως δημόσιο φορέα και τι ως ιδιωτικό για να αποφύγουμε την κερδοσκοπία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει αντί, ε, αντί για τις ε, κυρώσεις αυτές να έχουμε υψηλότερες. Δεν είναι δυνατόν να, έχουμε, να ζητάμε από κάποιον να πληρώνει σε 60 μέρες και από κάποιον άλλον συναλλασσόμενο να πληρώνει σε 30 μέρες. Δεν είναι ηθικό κατά τη γνώμη μου. Θεωρώ λοιπόν ότι οι καταποκοπήν ναι, κυρώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σωστές διότι ε, μιλάμε απλούστατα για το κόστος διεκπαιρέωσης και την κάλυψή του. Ε, εγώ θα πρότεινα να υπάρχει μία κλιμακωτή ε, κύρωση αναλόγως δηλαδή αν πρόκειται για ένα μικρό ποσό γράφουμε ένα γράμμα εάν είναι υψηλότερο το ποσό ορίζουμε ένα δικηγόρο και δεν είναι σωστό να έχουμε καταποκοπή αποκοπή π.χ χίλια ευρώ. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση αναλόγως με το ύψος της ε, κάθε απαιτήσεως. Και τέλος, η πρώτη μου τροπολογία αναφέρεται στις κυρώσεις. Πιστεύω ότι ο στόχος μας δεν είναι να εισπράξουμε τα 5 ευρώ. Νομίζω ότι για απαιτήσει πέραν των 5 ευρώ δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, με αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Και αυτό επειδή σήμερα υπάρχει ένα όριο 5 ευρώ και όταν πρόκειται μόνο για 5 ευρώ, ε, τότε δεν επιβάλλονται, δεν προστίθενται τόκοι καθυστέρησης στο 5 ευρώ, μόνο σε υψηλότερα ποσά. Ο νέος όμως κανονισμός ε, καταργεί αυτό το όριο. Εγώ θα ήθελα όμως αυτό το όριο να διατηρηθεί, διότι πιστεύω ότι διαφορετικά αυτό το πρόβλημα δεν θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Και πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολλές φορές ε, κερδοσκοπική στάση των ε, ε, δημοσίων εταιριών που περιμένουν οι υπεύθυνοι τους να συσσωρευτεί ένα μεγαλύτερο ποσό και δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν νωρίτερα. Finally, Mr. Last but not least, uh, I hope... Αυτό το οποίο δεν είδα είναι ε, η θέση των ε, τραπεζών. Στηρίζουμε τις ε, τράπεζες. Θέλουμε να περιορίσουμε την, υπερβολική χρηματοδότηση. Εάν λοιπόν αργούν τα βάλουν τις πληρωμές τους θα πρέπει και αυτοί να υφίστανται κυρώσεις. Αν πληρώνουν εγκαίρως τότε όλα πάνε καλά, δεν μας ενδιαφέρει. Απλούστατα μιλάμε για τον δημόσιο τομέα, για επιχειρήσεις που είναι κακοπληρωτές και καλό θα ήταν να μην πληρώνει κανείς μόνο κάποιο ευξημένο επιτόκιο αλλά και μία κύρωση. Ε, ελπίζω ότι οι θα μάθουν έτσι και θα μπορέσουμε να βρούμε μία λύση ε, για τις ε, πλεονασματικές αυτές πληρωμές ε, διότι ε, διαφορετικά οι εταιρείε ας χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες και ας καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους εν Αυτός είναι ο στόχος της τροπολογίας μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για μερικά πολύ χρήσιμα στοιχεία και ζητάω τώρα από την κυρία Μπρίνκμαν και μετά τον κύριο Μπράιν ε, αλλά προτού μιλήσει η κυρία Μπρίγκμαντ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν κοιτάξετε ε, τη λεπτομερή μελέτη των επιπτώσεων θα δείτε ότι ένα από, τα προβλήματα είναι η εναρμόνιση και αυτά όλα αναφέρονται ε, την μελέτη των επιπτώσεων. Άρα είναι ένα θέμα που έχει εξεταστεί εκτενώς σαν δυνατή και εφικτή εναλλακτική λύση οπότε καλό θα ήταν να το ξανακοιτάξουμε προτού αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Ε, καλό θα ήταν οι συγητές και οι σκιώδεις να τα ξανακοιτάξουν. Αλλά κύριε Μπρίνκμαν, θέλετε να μας πείτε ε, ποιες από τις τροπολογίες ε, θεωρείτε αποδεκτές και ποιες νομίζετε ότι είναι προβληματικές. Η κυρία Μπρίνκμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή στην ανάλυση των επιπτώσεων είχε εξετάσει αυτή την εναρμόνιση των προθεσμιών πληρωμής μεταξύ επιχειρήσεων και είχαμε καταλήξει στο ε, τελείως ε, αντίθετο συμπέρασμα. Με ακούτε. Λοιπόν, η Επιτροπή είχε καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα από την συνένεση η οποία, στην οποία καταλήγουν οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, απογοητεύουμε με μία, για μία τέτοια έκβαση διότι όλοι θέλουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως όσον αφορά την ανάλυση των μέσων για να επιτευχθούν οι στόχοι αλλά αντιλαμβάνουμε ότι διαφορετική είναι η ανάλυση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τι ορισμένες πολιτικές ομάδες που εξεφράστηκαν. Είναι όπως είπα απογοήτευση διότι στην τωρινή οικονομική κρίση η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι δύσκολη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό θεωρούμε ότι η εναρμόνωση ε, των ε, προθεσμιών πληρωμής μεταξύ ε, επιχειρήσεων θα διευκολύνει τη διακίνηση μεταξύ επιχειρήσεων και δεν θα χρειάζονται ε, και αν δεν έχουν αυτά τα χρήματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να πληρώσουν τις μεγαλύτερες ε, θα στραφούν προς τις τράπεζες οι οποίες σε αυτό το, περίοδο δεν είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν. Άρα έτσι δεν θα επιλύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι όντως ουσιαστικό για την καθυστέρηση των πιστωτών. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα ιδίως σε ορισμένους τομείς αλλά μην ξεχνάμε την μεγάλη πραγματικότητα των επιχειρήσεων οι οποίες χαίρουν από αυτό, αυτές τις πιστώσεις και θα μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν. Μας απογοητεύει λοιπόν αυτή η κατεύθυνση γιατί πιστεύουμε ότι όλοι θέλουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ήθελα να σας πω όσον αφορά για την μελέτη των επιπτώσεων ε, αναφέρουμε εκτενώς τα υπέρ και τα κατά και ε, εμείς θεωρήσαμε ότι ε, κάτι τέτοιο θα ήταν ε, μάλλον δυσμενές και όχι θετικό αλλά προφανώς δεν συμφωνείτε με τις ε, διαπιστώσεις μας. Επιπλέον υπάρχει το θέμα της εναρμονίσεως των προθεσμιών πληρωμών για, ε, από το δημόσιο, διότι εκεί ε, όντως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξασχίσουν καμία δυνατότητα πιέσεως και το δημόσιο ε, βρίσκεται σε τελείως διαφορετική θέση από τον ιδιωτικό τομέα όπως το είπαν άλλωστε ορισμένοι από εσάς και ε, το να μειωθεί η περίοδος πληρωμής στις 30 μέρες μας φαίνεται ε, ουσιαστικό. Δεν νομίζουμε ότι είναι λανθασμένο. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ε, εξέλιξη θετική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα απογοητευτούμε αν δούμε ότι και στο σημείο αυτό η πρόταση θα καταλήξει σε 60 ή και περισσότερες μέρες. Διότι αυτό νομίζω ότι θα απογοητευτούμε διαπραγματεύσει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και λήψη ε, χρόνου. Θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτά τα δύο στοιχεία. Η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας και είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε του τους καλύτερους συμβιβασμούς που μπορούν να σας βοηθήσουν και να μπορέσουν συγχρόνω να σταθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και κυρία Μπράιν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν συμβαίνει πολύ συχνά το να συμφωνεί κανείς απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λιγότερο με το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα το, ας το πω έτσι, την ανησυχία, το μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την παρέκκληση που σημειώνεται σε σχέση με την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, σε σχέση με τη γενική ιδέα. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Τον εναρμονισμό των προθεσμιών μεταξύ επιχειρήσεων που λεπτομερώς μελετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάλυση επιπτώσεων που έκανε και απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε επειδή ήταν μια κακή λύση αυτή. Παρακαλώ λοιπόν να το σκεφτείτε αυτό και να το στοχαστείτε γιατί θα ήταν πάρα πολύ βαρύ λάθος να επιμείνει το Κοινοβούλιο σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει πολύ νόημα οικονομικά. Μπορεί να φαίνεται εκ προημίου ότι ίσως επιλύονται προβλήματα. Όμως η αλήθεια είναι ότι πολλά περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται. Τόσα πολλά προβλήματα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απέρριψε και δεν την συμπεριέλαβε στην αρχική της πρόταση αυτή την εναλλακτική λύση. Και στην ανάλυση επιπτώσεων αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιους λόγους την απέρριψε. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν να λάβετε υπόψη παρακαλώ να είσαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ ε, επιφυλακτικοί για τον εναρμονισμό προθεσμιών μεταξύ επιχειρήσεων. Και εδώ έχουμε και την αντίθεση και του Συμβουλίου. Και εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το σημείο. Δεύτερο, συμμεριζόμαστε το ότι ο δημόσιος τομέας εννοείται ως διοίκηση, δημόσια διοίκηση, δημόσιες αρχές και που πρέπει οι κρατικές αρχές να έχουν κάποια όρια να χαλιναγωγηθούν για να μην υπάρξει κατάχρηση εξουσιών. Και συμφωνούμε σε αυτή την περίπτωση γενικά ως προθεσμία με κάποιες εξαιρέσεις που ζητήθηκε εξάλλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η προθεσμία είναι 30 ημερών, έτσι. Μετά στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε μια άλλη παρέκκληση που εισήχθη στο Κοινοβούλιο, διότι ανησυχούμε πολύ για αυτό το θέμα, με τη διεύρυνση του πεδίου, του τομέα, του τι καθορίζεται δηλαδή ως δημόσιος τομέας. Αυξήθηκε, επεκτάθηκε στις προτάσεις που υποβλήθηκαν μέχρι σημείου να συμπεριληφθεί και ένα δημόσιο τομέα πολύ ευρύτερος. Όσο περισσότερο διευρύνουμε όμως τον τομέα του δημοσίου ως έννοια, τόσο περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανταγωνισμό με ιδιωτικές επιχειρήσεις υπάρχουν και χρειάζονται για την ε, δραστηριοποίησή τους ισότιμο πλαίσιο ευκαιριών και όρων και προϋποθέσεων. Όταν διευρύνουμε το πλαίσιο, έχει αυτό αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την πιο αυστηρή αντιμετώπιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Δημιουργούνται δυσκολίες και γι' αυτό λοιπόν το Συμβούλιο είναι αρκετά αντίθετο, θα έλεγα αντίθετο απόλυτα στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Πιστεύουμε ότι το πλαίσιο του δημόσιου τομέα, όπως είχε καθοριστεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η σωστή λύση. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο, σε ένα από τα θέματα για τα οποία έγινε λόγος εδώ, για τις κυρώσεις ή τιμωρίες. Σε σχέση με το άρθρο 5, σημείο 5, το ότι δηλαδή το Συμβούλιο απορρίπτει κάθετα αυτές τις προτάσεις εμείς θεωρούμε σε σχέση με το Συμβούλιο ότι αυτό το 5% είναι ένα ποσό δυσανάλογο, απόλυτα δυσανάλογο και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Προβλήματα επειδή εισάγεται εδώ ως δέκτης, αποδέκτης της υποστήριξης ε, βοήθειας αυτής, αποδέκτης της κύρωσης διορθώνει ο μιλητής <clears throat> σε σχέση με τον την επιβαλόμενη ποινή. Υπάρχει η αντιστάθμιση λοιπόν, υπεραντιστάθμιση που μπορεί να προκληθεί. Αυτή η υπεραντιστάθμιση μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσεις τεράστιες. Ποτέ σε κανένα κράτος οι κυρώσεις δεν είναι ε, ευεργετικές σε εκείνους που τους επιβάλλονται. Οι κυρώσεις είναι ευεργετικές για το κράτος μόνο, για τον κρατικό κορβανά. Και εδώ εισάγεται μια νομική έννοια στρεβλή θα έλεγα που δημιουργεί στρεβλώσεις και είναι προβληματική και αυτό προφανώς που πρέπει να κάνουμε είναι να νομοθετήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγουμε προβλήματα και σήμερα και στο μέλλον και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ότι το Συμβούλιο βρίσκεται κοντά πολύ πιο κοντά στις αρχικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτός από το θέμα της κύρωσης του 5%. Στα υπόλοιπα είμαστε, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο Συμβούλιο στις αρχικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα θέλαμε αν είναι δυνατόν η Ευρωβουλή να αναθεωρήσει, να ξαναδεί τη θέση της και να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με αυτές τις θέσεις. Εγώ έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια προς την κυρία Βάιλερ και κατανοώ την τεράστια δυσκολία που συνεπάγεται για αυτήν το να αντιμετωπίσει αυτό το έργο, για να αντιμετωπίσει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι πολύ σύνθετο και ακαθόδες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω τις θέσεις του Συμβουλή. Δεν θέλω να ξανανοίξουμε νέο γύρο συζητήσεων. Πρόκειται για κάτι σημαντικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να ξεκινήσω νέα συζήτηση, αλλά με κάθε σεβασμό προς ε, την Επιτροπή δεν έχουμε καταλάβει την άποψη της Επιτροπής. Ο στόχος μας είναι κοινός. Διευκόλυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε τι μας λέτε για τις 30 ημέρες. Δεν καταλαβαίνουμε τι εννοείτε όταν μιλάτε για τους περιορισμούς. Τι ακριβώς είναι αυτό που σας απαγοήτευσε μήπως ε, να κοιτάξετε τις σελίδες 29, 30 και 31 της ε, ανάλυσης αντικτύπου και θα δείτε γιατί αποφάσισε η Επιτροπή να μην προτείνει πλήρη εναρμόνιση. Ίσως λοιπόν οι συνάδελφοι που συμφωνούν μαζί σας θα έπρεπε να διαβάσουν αυτό το κομμάτι. Μπορεί να διαφωνείτε βεβαίως, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα επιχειρήματά σας είναι βάσιμα αν λάβουμε ως βάση αυτή την καλή κατά τη γνώμη μου εκτίμηση επιπτώσεων. Και να πω ότι στην αρχή της διαδικασίας εξετάσαμε εντελεχώς την εκτίμηση επιπτώσεων. Υπάρχουν ε, αρκετοί συνάδελφοι που προτιμούν ε, να μην συμφωνήσουν με αυτή, πολύ καλά, αλλά θα έπρεπε να διπλοτσεκάρουν τέτοιου είδους διαφωνίες. Αυτό το λέω ειδικά και για την κυρία Χάνσλικ, η οποία νομίζω ότι ήταν η βασική υπεύθυνη για αυτή την απόφαση και αυτή ήταν η ουδέτερη στάση μου ως πρόεδρου. Κύριε Ντιόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Για δεύτερη φορά μας λέτε να εξετάσουμε την μελέτη επιπτώσεων. Μα ειλικρινά πιστεύετε ότι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ως κοιόδης εισηγητής χωρίς να διαβάσουμε τα έγγραφα. Φυσικά και τα διαβάσαμε, αλλά πέρα από αυτά μιλήσαμε και επιχειρηματίες με εκπροσώπους μεμονωμένων επιχειρήσεων. Και αν το είχατε κάνει και εσείς κύριε Πρόεδρε θα είχατε διαπιστώσει ότι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και ότι επιθυμούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς αυτές τις προτάσεις. Όχι γιατί δεν έχουμε διαβάσει την εκτίμηση επιπτώσεων, αλλά συζητήσαμε και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που το κάνατε. Ναι, και προκαταλάβατε και την δική μου υπόδειξη σχετικά. Το δεύτερο θέμα τώρα, η νομική θέση της πρότασης. Αν συμφωνούν οι συντονίστες, θα ήθελα να ζητήσουμε από τον νομικό μας σύμβουλο να έρθει στην συνάντηση των συντονιστών και να κάνουμε κάποια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά. Κυρία Βάιλεν, μήπως μπορούμε να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Ευχαριστώ. Σε κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια να απαντήσω πρώτα. Καταρχήν για την τελευταία παρατήρηση Γνωρίζω ότι οι συνάδελφοί μου, σκιώδεις εισηγητές, φυσικά έχουν διαβάσει όλα τα έγγραφα. Κατά κανόνα ήταν όλοι παρόντες όταν συζητούσαμε με εκπροσώπους ενώσεων και συλλόγων και γνωρίζουν όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, όλα τα υπέρ και όλα τα κατά. Και κάποτε πρέπει φυσικά να ληφθεί μια πολιτική απόφαση από μας. Και τώρα έρχομαι στο πρώτο σημείο λοιπόν, στο Συμβούλιο σχετικά. Κατανοώ ότι το Συμβούλιο έχει απογοητευθεί, νιώθει απογοήτευση, αλλά αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία και διεργασία με πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες και πολιτικές ομάδες που εμπλέκονται. Και αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Και πρέπει να πω δόξα τω Θεώ. Δεν υπάρχει καμιά μόνη της κοινοβουλευτική ομάδα που να μπορεί να επιτύχει την θέσπιση ενός νομοθετήματος. Από κοινού πρέπει να τα καταφέρουμε. Από κοινού μόνο μπορούμε να τα καταφέρουμε. 27 κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ των ομάδων. Και δεν είναι απλή υπόθεση να μπορεί κανείς να συνεννοηθεί εύκολα για αυτά τα θέματα όπω και εμεί και οι σκιώδει εισηγητέ. Αλλά έχουμε και διαφορετικά συμφέροντα εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο από το Συμβούλιο. Έχουμε και διαφορετικά εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τα κράτη-μέλη μα ούτω ή άλλω. Είναι λοιπόν μια δημοκρατική διαδικασία και διαργασία αυτή. Και πρέπει να μπορεί κανεί να, να δεχτεί και αλλαγέ και μεταβολέ. Και εγώ ίδια και το μεγαλύτερο μέρο τη ομάδα μου θα ήταν υπέρ τη δια, διατήρηση τη συμβατική ελευθερία. Και μέσα στο πλαίσιο της συμβατικής ελευθερίας κάποιους κανόνες που θα έπρεπε να θεσπίσουμε. Βλέπω και αναγνωρίζω ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί όμως πλειοψηφία με μια τέτοια θέση και είμαι πρόθυμη να υιοθετήσω διαφορετική θέση. Κυρία Μπρίνκμαν, πιστεύω ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν ρόλο υποδείγματος και παραδείγματος. Θέλω να απευθύνω έκκληση να μην επαναλάβουμε κάτι το οποίο ε, από το Δεκέμβριο έχει αφαιρεθεί από το τραπέζι, δηλαδή το 5% των χειρόσεων. Ευθύ εξ αρχή, ήδη στην πρώτη συζήτηση σε αυτή την Ευρωβουλή, είμαστε όλοι τη γνώμη και δεν άκουσα κάποια διαφορετική άποψη ότι το 5% είναι υπερβολικά υψηλό ποσό. Και μετά από ένα εξάμεινο συζητήσεων δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το σημείο του 5%. Το 5% ποτέ δεν είχε τεθεί υπό Αν παίρναμε 2% όπως πρότεινα εγώ η ίδια ή εναλλακτικά όχι ε, ε, μια, ε, ε, όχι τίποτα άλλο παρά μια αύξηση των τόκων υπερημερίας. Για, θα ήταν κάποια διαφορετική ας το πούμε αυτή η εναλλακτική εφαρμογή. Αλλά πάλι κύρωση. Γιατί χωρίς κανόνες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Ξέρουμε το νομοθέτημα του 2000 και αυτό δεν επαρκούσε. Θέλω πάλι να δραχθώ της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία της Ευρωβουλής και να απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους την ιδιαίτερη αυστηροποίηση, αυστηροποίηση το ιδιαίτερα αυστηρότερο πλαίσιο που δημιούργησε η νομική επιτροπή να μην το υποβαθμίζουμε. Δεν θα ρυθμίσει όλα τα προβλήματα βέβαια, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά εμπλουτίζει το πλαίσιο του νομοθετήματος και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν θέλουμε να έχουμε ένα νέο νομοθέτημα το οποίο και απευθύνουμε έκκληση στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα νόμο όπως στη Γαλλία όπου εκατοντάδες εξαιρέσεων συμπεριλαμβάνονται και, συμπεριλαμβάνονται και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται τελικά. Και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι το θεωρούν και πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο λέει είναι μη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Αν θέλουμε να κάνουμε μια, ένα ε, λειτουργικό νομοθέτημα και βιώσιμο νομοθέτημα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς γραφειοκρατική επιβάρυνση. Απευθύνω έκκληση να κρατήσουμε και να αντέξουμε μέχρι τέλους και να μην δεχθούμε επιρροή όποιων συλλόγων και ενώσεων όποιε προθέσεις, καλές προθέσεις μπορεί να έχουν να κάνουμε εξαιρεσει για αυτού και για αυτές. Το λέω αυτό και προσωπικά διότι γνωρίζω τη δημιουργικότητα των συναδέλφων μου και το ζήσαμε και το βιώσαμε στη φιλελεύθερη ομάδα τρεις διαφορετικοί συνάδελφοι με τρεις διαφορετικές απόψει. Και στι άλλε ομάδε υπάρχουν ε, τέτοιε ε, διαφορές. Ε, συγγνώμη, είσαστε οι πράσινοι που ήταν πάντα, συνεπεί στη θέση της. Οι υπόλοιποι πρέπει να πω ότι πολλές φορές άλλαζαν θέση. Πρέπει να έχουμε το θάρρος μέχρι τέλους να παραμείνουμε πιστοί και συνεπεί στην απόφασή μας. Να μην ακολουθήσουμε κάποιες παρεκκλήσει νομικέ. Είναι πολιτική απόφαση. Αν θα υιοθετήσουμε και θα ακολουθήσουμε την πορεία της συμβατικής ελευθερίας νέου. Πιθαν... Δυνατό είναι αν το θέλουμε, αλλά το θέμα είναι αν ε, το θέλουμε όλοι. Το ίδιο είναι ότι θα μπορούσε κανείς να εισαγάγει κυρώσει και ποινές. Αν το θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά αν δεν θέλουμε να το κάνουμε, ας έχουμε το θάρρος να πούμε όχι, έχουμε μια άλλη εναλλακτική λύση, κάποια άλλη πορεία θέλουμε να ακολουθηθεί. Δεν θέλω να ακολουθήσουμε μια, ας το πω έτσι, ομφαλοσκόπηση νομικίστικη και να λέμε κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γιατί νομικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εφόσον πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ρύθμιση και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ας είμαστε συνεπείς σε μια τέτοια θέση. Και αν πιστεύουμε ότι οι τόκοι υπερημερίας πρέπει να αυξηθούν σε καθυστέρηση, καθυστέρηση πληρωμών πρέπει να είμαστε, συμ, συνε, να, να είμαστε με συνεκτικοί και συνεπείς. Διότι για οποιαδήποτε άλλα μέσα για την επίτευξη του στόχου το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα συνεκτικό νομοπλαίσιο. Να μην έχουμε ένα νόμο που ίσως για τρεις μήνες μετά από την έγκρισή του θα καταλήξει σε κάποια δικαστήρια με προσφυγές και με κάποιες ε, μομφές. Δεν είναι αυτό το οποίο είναι ε, υπέρ του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν ας καταφέρουμε μέσω του Στρασβούργου μέχρι το Στρασβούργο να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα αποτελεσματικό που μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Τώρα αν ο ένας ή η άλλη συνάδελφος δεν θέλει να ακολουθήσει αυτή την πορεία τότε αυτή είναι η δημοκρατική μας ζωή πρέπει να το δεχτούμε αυτό αλλά πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε μια ευρεία πλειοψηφία και για τις ε, περίπλοκες ε, διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε, Μπάρμπαρα Βάιλερ για την ηγετική στάση που έπαιξε στη συζήτηση αυτού του φακέλου αλλά και όλους για την βοήθειά τους. Ψηφοφορία μάλλον θα έχουμε 28 Απριλίου. Είχαμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων σήμερα και νομίζω ότι θα έχουμε μια ακόμη και επίσης νομίζω και σίγουρα θα το κάνει η κυρία Βάιλερ με τους κοιόδης εισηγητές ότι πρέπει να εξετάσουμε το τι θα κάνουμε και με το Συμβούλιο. Γιατί σίγουρα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εφόσον μιλάμε και για έναρξη ισχύων 20 ημέρες μετά, είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη. Βεβαίω οι συνάδελφοι θα αποφασίσουν αν θέλουμε να επιβραδύνουμε τη διαδικασία για αρκετού μήνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουν οι συγκεκριτέ ε, και η κυρία Βάιλερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα κλείσω τη συνεδρίαση και στις 6 θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα έχουμε την νομική υπηρεσία αλλά και την κυρία Βάις Κέρμπερ η οποία θα μας μιλήσει για την πρόταση της καθώς και για την πιθανότητα να έχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Επανερχόμαστε αύριο το πρωί στις 9 στην ίδια αίθουσα με τις εκθέσεις Grace καθώς και με την συνάντησή μας με τον κύριο Μόντι. Ευχαριστώ. Uh, Παρακαλώ, όποιος δεν έχει να κάνει με τους συντονιστές να φύγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Υπάρχει αρκετός χώρος έξω για να συνεχίσετε τις συζητήσεις.